Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. συνεχίζουμε. Προφορική ερώτηση για την ανάπτυξη δορυφορική τεχνολογία για να οι επεκτάτα ζητήματα παγκόσμια παρακολούθηση πτήσεων. Τελεία. Αυτό είναι ο τίτλο. Ο κύριος Κράμερ πρώτος. Mr. Kramer, you have the floor. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμη συνάδελφη, κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόμα τη Επιτροπή Μεταφορών θα ήθελα να καταθέσω προφορική ερώτηση με θέμα ανάπτυξη δορυφορική